για την παρατήρηση και την πληροφορία που μου δώσατε. Έλαβα από την ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος ε, και από την ομάδα της Ενωτικής Αριστεράς ε, τήσει ε, για διορισμούς ε, στις επιτροπές και τις κοινωνικές ελπισοπίες. Ο κατάλογος των ε, διορισμών θα συμπεριληφθεί στα πρακτικά της Συνόδου. Εάν δεν έχει υπάρχει καμία ένσταση, τότε αυτές οι... Αυτοί οι διορισμοί θα θεωρούν εγκεκριμένοι. Έχετε λοιπόν τα ονόματα στον φάκελό σας τώρα. Η υπογραφή των νομοθετικών